Επιτροπή, αντίστοιχα θα τύχουν αντιμετώπιση από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και προσβλέπω στην μελλοντική μας συνεργασία τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγη συζήτηση. ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Τετάρτη.